Καλώς ορίσατε. Ελπίζω να είστε ξεκούραστοι, φρέσκοι, έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις 8.000 τροπολογίες που μας αναμένουν. Και να ξεκινήσουμε λοιπόν τη σημερινή συνεδρίαση με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν υπάρχουν ενστάσεις, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Να σας ανακοινώσω επίσης ότι υπάρχει διερμηνία σε όλες τις γλώσσες για τη σημερινή συνεδρίαση. Σημεία υπαριθμών 2. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 18ης και 19ης Ιουνίου, της 25ης Ιουνίου και 9ης και 10ης Ιουλίου 2012. Αν δεν υπάρχουν σχόλια μέχρι το πέρας της συνεδρίασης, θα θεωρούμε ότι εγκρίθηκαν και τα πρακτικά. Να σας ενημερώσω επίσης ότι η σημερινή συνεδρίαση μεταδίδεται μέσω webstream. Και να σας πω επίσης ότι η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου με ενημέρωσε ότι ετοιμάζει μία έκθεση πρωτοβουλίας για τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, για την οποία θα ψηφίσει στις 10 Οκτωβρίου. Επειδή ο αυτό δεν επιτρέπει στην Επιτροπή μας να ε, ετοιμάσει σχετική γνωμοδότηση. Σας προτείνω να παρουσιάσετε τροπολογίες απευθείας στην Γραμματεία της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου πριν από τις 19 Σεπτεμβρίου. Να σας ενημερώσω επίσης ότι ο μεγάλος όγκος των τροπολογιών που σας διανεμήθηκε δεν θα διανεμηθεί σε άλλα αντίγραφα, Γι' αυτό λοιπόν κρατήστε σε αυτές τις τροπολογίες. Και αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε στο σημείο υπαριθμών 4, Γενικός Προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013. Η Εστέρ Ντελάνγκε είναι εδώ μαζί μας να σας πω ότι το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του για τον προπολογισμό για το 2013 μόλις πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές στις 24 ε, Ιουλίου και επιβεβαίωσε ότι έχει πρόθεση να ζητήσει περικοπές σε αρκετές γραμμές του προπολογισμού της κοινή γεωργικής πολιτικής όπως για παράδειγμα τις δράσεις προώθησης και τα προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική η σημερινή ψηφοφορία θα ψηφίσουμε επί 35 τροπολογιών για τον προπολογισμό για το 2013. Να υπενθυμίσω επίσης στους συναδέλφους ότι στην επόμενη συνεδρίαση της 18 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε για τη γνωμοδότηση που συνοδεύει τις ε, τροπολογίες μας. προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι η 4η Σεπτεμβρίου, δηλαδή αύριο στις 12 το μεσημέρι. Να ε, χαιρετήσω και το Γενικό Διευθυντή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι εδώ μαζί μας. Δεν ξέρω αν η κυρία Ντελάνγκε θέλει το λόγο, αλλιώς μπορούμε να περάσουμε απευθεία στην ψηφοφορία. Να ψηφίσουμε λοιπόν. Αν συμφωνείτε, ε, για να ολοκληρώσουμε πιο γρήγορα θα ψηφίσουμε δυνατά ο ισχυρός. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν. Ξεκινούμε με την τροπολογία 5.200. Υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι πρέπει να το επαληθεύσουμε. Απορρίπτεται νομίζω. Αποχές. Ωραία. Απορρίπτεται. 52-19. Άρχεται η ψηφοφορία. Υπέρ. Κατά. Κατά, Λουίς. Γιατί 52-19. Ωραία. Αποχές. Απορρίπτεται. 52-29. Υπέρ. Κατά. Κατά αποχές εγκρίνεται. 52-18 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να επαληθεύσουμε την 52-18. Να ελέγξουμε λοιπόν αν υπάρχουν ε, οι κάρτες σας. Έχετε, ωραία. 52-18. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 52-23. Άρχεται η ψηφοφορία για την 52-23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Η Εγκρίνεται. 52-01 και η 52-17 είναι ταυτόσιμες υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 5202-5216 υπέρ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5203 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5226 52-26 υπέρ. Υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 52-19 υπέρ. Για την 52-19 υπέρ, κατά. Να κάνουμε μια παλήθευση. Για την 52-19, Μία γρήγορη επαλήθευση. Ψήφισαν όλοι. Απορρίπτεται. Πενήντα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 52-27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52-25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52-19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήταν μεγάλη διαφορά στα καποιο επαληθευση επαλήθευση. 52-24 τώρα. «52-19 για τις αποζημιώσεις για τα πουλερικά. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. κατά, αποχές, απορρίπτεται. «52-24 υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 52-32 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 52-31 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 52-34 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 52-20 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται θα έλεγα, να κάνουμε μια παλήθευση. 52-20. Ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι για τον καπνό. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 15 κατά 11 υπέρ. Απορρίπτεται λοιπόν. 52-04 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 52-21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 52-13 ε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 52-07 υπέρ, 5209, συγγνώμη, 5209 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα 5207 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 5208 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 5233 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 5206 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5211 υπέρ. Κατά. Αποχές 5212 Υπέρ. Κατά. Αποχές. 5205 Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τέλος, η 52-22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ωραία, σας ευχαριστώ. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε την Εστέρ Δελάνγκη για τη δουλειά της και προχωρούμε. Να σας υπενθυμίσω λοιπόν Πέρας κατάθεση τροπολογιών 4 Σεπτεμβρίου 2012 για το σχέδιο της νομοδότησης. Περνάμε τώρα στο σημείο 5. Την προσοχή σας λίγο παρακαλώ. Είμαστε στην πρώτη πράξη κατεξουσιοδότηση για το γεωργικό τομέα, για το γαλακτοκομικό τομέα, ε, του οποίου προσφάτως εγκρίναμε τη δέσμη μέτρων. Να υπενθυμίσω ότι η Επιτροπή παρουσίασε την πρώτη πράξη κατά που θέλει να καθορίσει κανόνες που σχετίζονται με την αναγνώριση των οργανώσεων ε, παραγωγών που δραστηριοποιούνται διαμεθοριακώς και τις ε, διεθνείς οργανώσεις παραγωγών, καθώς επίσης και την ε, σύσταση και τις προϋποθέσεις διοικητικής συνδρομής που θα πρέπει να παρέχεται σε περίπτωση τέτοιας διαμεθοριακές συνεργασίες και επίσης τον ε, τομέα του γάλακτος, ε, το οποίο καλύπτεται από διαπραγματεύσεις των οργανώσεων των παραγωγών και ε, όσων κάνουν μεταποίηση γάλακτος. Βάσει του άρθρου 290 της Συνθήκης της Λισαβόνας, αυτή η πράξη κατά εξουσιοδότηση μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή μόνο όταν δεν έχει ενστάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός συγκεκριμένη προθεσμίας. Αυτό είναι ο ρόλο που έχουμε δώσει σε αυτέ τι πράξει κατά εξουσιοδότηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ζήτησε από το Κοινοβούλιο να εκφράσει την άποψή του με κατεπίγουσα διαδικασία ώστε να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ ε, η πράξη αυτή στις 3 Οκτωβρίου του 2012. Η επιστολή η οποία δικαιολογεί το κατεπήγον τα χαρακτήρα αυτής της πρότασης ε, σας έχει διανεμηθεί και καθορίσαμε ως προθεσμία για τις ενστάσεις μας ε, την 29η Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι. Επειδή δεν υπήρξε καμία ένσταση, καμία αντίρρηση, προτείνω λοιπόν να εγκριθεί η σύσταση μέσω ε, της ε, διαδικασίας αυτής της μη αντίρρησης στην πράξη κατεξουσιοδότηση. Βάσει λοιπόν του άρθρου 17α μπορούμε να παρουσιάσουμε τη συγκεκριμένη σύσταση στην επόμενη Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου, ε, όταν βέβαια φυσικά δώσουν την έγκρισή του ε, και η διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών. Αυτή είναι η πρότασή μου. Ποιο είναι λοιπόν αυτή, υπέρ αυτή τη επιλογή, να δώσουμε την έγκρισή μα, είστε όλοι υπέρ, υπάρχουν κάποιε στάσει. Όχι, ωραία, εγκρίνεται αυτή η πράξη κατά εξουσιοδότηση λοιπόν και θα ψηφιστεί στην επόμενη Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Ευχαριστώ πολύ του συναδέλφου. Και τώρα μια άλλη σύντομη ενημέρωση για το σημείο 6. Ενδιάμεση έκθεση εν ώψη της θετικής έκβασης της διαδικασίας έγκρισης του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, οι συζητήσεις για το μελλοντικό δημοσιονοϊκό πολιετές πλαίσιο είναι υψής σημασία σημασίας για την κοινή γεωργική πολιτική και τη διαδικασία μεταρρυθμίσεων την οποία συζητούμε επί του παρόντος. Η γνωμοδότησή μου βασίζεται στο γεγονός ότι υπάρχει άποψη του Κοινοβουλίου ε, στην έκθεση 28 Ιουνίου της Επιτροπής ΣΟΥΡΕ, καθώς επίσης και μία έκθεση της 23 Ιουνίου, η έκθεση ΝΤΕΣ. Και στις δύο περιπτώσεις σας υπενθυμίζω ότι το Κοινοβούλιο ζήτησε σαφέστατο ο προπολογισμός της κοινωνικής πολιτικής να παραμείνει τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με τον παρόντα προπολογισμό για το παρόν πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και αυτό με πραγματικούς όρου, και αυτή είναι και η θέση μας μέχρι και σήμερα. Όπως θα είδατε λοιπόν στο σχέδιο γνωμοδότησης που σας είχαμε παρουσιάσει πριν από τι καλοκαιρινές διακοπές, οι προτάσει της, Ευρωπαϊκής, της Επιτροπής μας Συγγνώμη, οι προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελούν σημαντική μείωση σε πραγματικού όρου για τον προπολογισμό τη κοινή γεωργική πολιτική. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ζητήσουμε αύξηση των ποσών για την δεύτερη κατηγορία, αν θέλουμε να ε, έχουμε τον ίδιο προπολογισμό σε πραγματικού όρου. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε πάγωμα του προπολογισμού και όχι περικοπή, όπω γίνεται αυτή τη στιγμή και μα προτείνεται. Μας ενημέρωσε επίσης το Συμβούλιο ότι οι χώρες που είναι καθαροί συνεισφορείς θέλουν να μειώσουν τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ κάποιες άλλες χώρες ε, ε, θέλουν να έχουμε πιο στοχευμένες δαπάνες η συνολική μείωση του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης βεβαίως θα έχει ε, επιπτώσεις και για τον προπολογισμό της κοινή γεωργικής πολιτικής. Η μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής ε, σημαίνει ότι θα πρέπει οι γεωργοί να κάνουν πολύ περισσότερα και αυτό το έχουμε δει και σε προτάσεις που καταθέσατε εσείς, καταθέσαμε όλοι εδώ στην ομάδα. Ζητάμε να υπάρχουν ε, περισσότερα δημόσια αγαθά, να τηρούνται καλύτερα πρότυπα πιο αυξημένα σε σχέση με τις ε, άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να επιτευχθεί με περικοπές στον προπολογισμό. Είμαι εν αναμονή λοιπόν των σχολείων σας και να σας επενθυμίσω ότι και για αυτή τη γνωμοδότηση θα πρέπει να κατατεθούν τροπολογίες μέχρι αύριο στις 4 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Να ξεκινήσει λοιπόν τώρα η συζήτηση. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος ο οποίος θέλει να λάβει το λόγο. Έχω ήδη την Έστερ Ντελάνγκε, τον Τζορτζ Λάιον και φυσικά ε, και οποιοδήποτε άλλο θέλει να σχολιάσει. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον Τζορτ Λάιον. Παρακαλώ. Ε, thank you. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ και για το σχέδιο γνωμοδότησης που μας έχετε υποβάλει στην Επιτροπή μας. Πολλά από αυτά που λέτε με βρίσκουν σύμφωνο. Όχι 100% βέβαια και δεν είμαι κατά 100% πεπισμένος ότι και η έκθεση Lion και η, έκθεση DES είναι σαφή σε σχέση με το τι ακριβώς θα πρέπει να σημαίνει ο προπολογισμό να μείνει στο επίπεδο του 2013. Χρειάζεται προσοχή στα θέματα αυτά. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για αυτά που θα πούμε για τις πολιετής δημοσιονομικές προοπτικές και την τελική απόλυξή τους. Είχαμε προτάσεις της Κομισιόν για τα θέματα αυτά και όπως είπατε σε πραγματικούς ε, όρους μιλάμε για 10% μείωση όταν σε άλλους τομείς υπάρχει απλώς πάγωμα ή ενδεχομένως και αύξηση. Αλλά δεν υπάρχει καμία άλλη περιοχή του προϋπολογισμού, κανένας άλλος τομέας που να περικόπτεται όσο η γεωργία. Η πρόταση της Κομισιόν αντιμετωπίστηκε ως σημείο αναφοράς και σημείο κίνησης στις διαπραγματεύσεις του Συμβουλίου. Γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή για το τι ακριβώς θα πούμε. Και η δική μου πρόταση θα ήταν αντί να ζητήσουμε να, επαναληφθεί, να επαναφερθεί ο προϋπολογισμός στο προηγούμενο επίπεδο σε πραγματικούς όρους, δηλαδή να υπάρξει αυτή η αύξηση κατά 30 δισεκατομμύρια ουσιαστικά στην πολυετή αυτή η περίοδο, νομίζω μια πιο πολιτικά λογική στάση για την Επιτροπή μας είναι να επισημάνουμε στο Κοινοβούλιο και να τονίσουμε ότι η γεωργία είναι ο μόνος τομέας ο οποίος βάσει των τωρινών προτάσεων θα υποστεί τέτοια σημαντική μείωση. Εάν πρόκειται να υπάρξουν λοιπόν μειώσει στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο φαίνεται να διαγράφεται ω μια πιθανότητα τουλάχιστον στο Συμβούλιο, δεν θα πρέπει η γεωργία να είναι το πρωτοθύμα αυτών των περικοπών. Οι περικοπές και οι εξοικονομήσεις θα πρέπει να προέλθουν από άλλους πολιτικούς τομείς. Είναι απαραίτητο λοιπόν να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα στο κοινοβούλιο μας που ίσως δεν έχουν καταλάβει ότι ήδη η Κομισιόν προτείνει σημαντικές περικοπές στις αγροτικές δαπάνες. Αν λοιπόν υπάρξουν περαιτέρω περικοπές στο συνολικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί θα πρέπει να αναζητηθούν άλλοι τομείς όπου θα υπάρξουν περικοπές και όχι μόνο η γεωργία. Ελπίζω λοιπόν θα κατατεθούν κάποιες τροπολογίες προς την κατα... κατεύθυνση αυτή και ελπίζω θα με υποστηρίξουν και οι συνάδελφοι. Είναι μια επιφυλακτική αλλά και σόφρον θέση της Επιτροπής μας πιστεύω αυτή είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε μια αξιοπιστία ως Επιτροπή Γεωργίας για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ, Τζόρτζ. Δίκιο έχεις, πιστεύω. Προσπαθήσουμε να λάβουμε υπόψη αυτές τις παρατηρήσεις που μου φαίνονται ιδιαίτερα εύστοχες, γιατί πράγματι η Γεωργία αυτή τη στιγμή είναι ο μόνος τομέας ο οποίος είναι στην κλίνη του προκούρου αυτή τη στιγμή και δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να σας συγχαρώ για την έκθεσή σας. Είναι σαφές από την έκθεση αυτή πώς η Κομισιόν έχει προσπαθήσει να καλοποιήσει τα στοιχεία στον προϋπολογισμό για να μας δώσει την εντύπωση ότι ο προϋπολογισμός της γεωργίας απλώς παγώνει όταν μειώνεται ουσιαστικά και σημαντικά. Και το να έχουμε και άλλα εργαλεία εκτός της κοινής αγροτικής πολιτικής, αυτό μπορεί να φαίνεται θετικό και ωραίο αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουν καθόλου χρηματοδότηση. Οπότε είναι εικονικό αυτό μονάχα το εγχείρημα της Κομισιόν σε σχέση με τη χρηματοδότηση άλλων τομέων της γεωργίας. Εγώ συμφωνώ με αυτά που λέει ο Τζόρτζ. Διάβασα την έκθεσή του προσεκτικά το καλοκαίρι, αλλά ενδιάμεσα έχουν γίνει πολλά πράγματα. Θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν ιδιαίτερα ανάλυφο και σαφέ σε όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου πόσο έντονε ήταν οι περικοπέ στη Γεωργία σε σχέση με άλλου τομεί και θέλω και αυτό να υπογραμμιστεί. Και σε σχέση με την επαναφορά των στοιχείων του προπολογισμού των αρχικών αριθμών και εδώ, George, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί πώς θα το διατυπώσουμε χωρίς να χάσουμε την διαπραγματευτική μας θέση, δεν θέλουμε να υποχωρήσουμε αμέσως. Χρειάζεται μια προσεκτική λοιπόν διατύπωση για το πώς πρέπει να διατηρηθούν τα κονδύλια αυτά. Δεν πρέπει εμείς να βάλουμε τον εαυτό μας εκτός παιδιάς και εκτός συζήτησης σε σχέση με τα κονδύλια του προϋπολογισμού. Κάτι που συζητήσαμε επίσης στην ομάδα μας ήταν το σημείο 7 που αναφέρεις που ζητάει ευκαμψία να μπορεί κανείς να διακινεί ποσά μεταξύ των δύο πυλώνων της κοινή αγροτικής πολιτικής. Αυτό σίγουρα είναι μια δυνατότητα που συζητείται για τη μελλοντική αγροτική πολιτική. Δεν θέλω λοιπόν να το βγάλω αυτό από το πλαίσιο αυτό, αλλά να τονίσω ότι και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη στο μυαλό μας όταν προχωρούμε σε μεταρρυθμίσεις, σε αποφάσεις για τη μεταρρυθμίση της ΚΑΠ, να έχουμε και αυτό στο μυαλό μας. Δεν θέλουμε λοιπόν να υποστηρίξουμε κάτι το οποίο στις τελικές αποφάσεις θα τροποποιηθεί τελείως. Αυτά λοιπόν ήθελα να πω και εγώ εξ ονόματος της ομάδας μου και ευχαριστώ και πάλι για την έκθεση με την οποία συμφωνώ σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ευχαριστώ Έστηρ, πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σεκεριάς και ο Αντιπρόεδρος και θα ήθελα να ακούσουμε από εκεί και πέρα τους υπολείπους αν έχουν να προσθέσουν κάτι. Rzeczywiście sytuacja Ευχαριστώ. Τα βλέπω τα πράγματα λίγο δύσκολα. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα που ασχολούμαστε με τα θέματα των πολιτικών δημοσιονομικών προοπτικών, νομίζω ότι έχουμε κρατήσει μια ιδιαίτερα εξισορροπημένη και μετριοπαθή στάση για τα κονδύλια. Ξέρουμε τις θέσεις των κρατών μελών, ξέρουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα οικονομικής κρίσης, ένα πρόβλημα υπερχρέωσης των κρατών μελών. Αλλά ίσως έχουμε ελαφρά την καρδία αποδεχθεί πολλές περικοπές στον προϋπολογισμό μας. Για όλα αυτά. Η κατάσταση είναι πράγματι πολύπλοκη. Τίθεται το ερώτημα. Πώς θα αντιδράσουν και οι γεωργοί στις αποφάσεις αυτές. Βλέπουν ότι θα περιοριστεί το εισόδημά τους. Επίσης, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένας προϋπολογισμός αναπτυξιακό ο οποίος έχει αντικυκλικό αποτέλεσμα σε σχέση με την κρίση και αυτό πρέπει να το τονίσουμε μέσα στα πλαίσια της συζήτησης η μεταρρύθμιση της κοινή αγροτική πολιτικής θα φέρει θετικά αποτελέσματα σε όλους και στους καθαρούς συνεισφορεί και στους καθαρούς αποδέκτες κονδυλίων. Κάτι ακόμα. Εγώ μπορώ να φανταστώ <clears throat> πού θα γίνουν οι περικοπές, όχι στον πρώτο πυλώνα. Γιατί ο πρώτος πυλώνας ουσιαστικά εξασφαλίζει μία ροή κονδυλίων στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό φαντάζομαι ότι οι περικοπές θα λάβουν χώρα στον δεύτερο πυλώνα, γιατί ο δεύτερος πυλώνας ουσιαστικά υποστηρίζει την αντιμετώπιση προβλημάτων του περιβάλλοντος, υποστηρίζει μια οικολογική προσέγγιση. Είναι ο τομέας αυτός ο οποίος θα πρέπει να δώσει και μια ιδιαίτερη υποστήριξη στα νέα κράτη-μέλη. Η ισορροπία λοιπόν μεταξύ των δύο πυλώνων δεν θα πρέπει να τροποποιηθεί. Φυσικά πρέπει να έχουμε μια εξισορροπημένη γνωμοδότηση, αλλά θα πρέπει να είμαστε σαφείς. Γιατί θα πρέπει να τονίσουμε ποιες είναι οι προσδοκίες των γεωργών ενώπιον της παγκόσμιας οικονομικής κατάστασης. Γι' αυτό θα πρέπει να έχει μια τέτοια σαφήνεια η γνωμοδότησή μας και σύμφωνα με τους προλαλήσαντες θα ήθελα να είναι πιο ίσως έντονη η διατύπωση στη γνωμοδότησή μας. Αυτός είναι ο νόμος, ο λόγος ύπαρξής μας. Θα μας ρωτήσουν τι ρόλο παίξατε στη διαμόρφωση αυτής της απόφασης. Ευχαριστώ. Γεια και Μποβέ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον ε, Πρόεδρο και εισηγητή για αυτή τη γνωμοδότηση. Είχαμε πάρει διάφορες ε, ανακοινώσεις από την Επιτροπή και δια του στόματος του ιδίου του Επιτρόπου για τα θέματα αυτά. Αλλά εμείς εκπροσωπούμε εδώ τους γεωργούς. Οι γεωργοί δεν ενδιαφέρονται για αυτά τα οποία είναι στις εφημερίδες ή στις δηλώσεις των Επιτρόπων. Τους ενδιαφέρει τι ακριβώς θα πάρουν σε επίπεδο επιδοτήσεων στην πράξη. Αν θα είναι περισσότερα ή λιγότερα τα χρήματα αυτά. Η Κομισιόν, όπως ελέγχθη, μπορεί θαυμάσια να παρουσιάζει τα μαύρα ως άσπρα και να καλοπίζει τις πραγματικότητες. Αλλά τώρα έρχεται <clears throat> στο σημείο που εμείς θα πρέπει να, να δούμε τα συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία. Λοιπόν, τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται δύσκολα. Εγώ δεν με ενδιαφέρει πώς θα τα ονοματίσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Για μένα το σημαντικό είναι να παραμείνουμε στο ίδιο επίπεδο ονομαστικά τουλάχιστον από ότι στον προηγούμενο, ε, στην προηγούμενη περίοδο δημοσιονομικών προοπτικών. Πώς θέλετε να το διατυπώσετε αυτό δεν με ενδιαφέρει. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει να εξασφαλίσουμε τη διατήρηση του συνολικού ποσού και αν υπάρχουν τώρα αποχρόντες λόγοι, αν υπάρχουν λόγοι που μας υποβάλλουν, επιβάλλουν μια διαφορετική αντιμετώπιση, αν λοιπόν υπάρχει κάτι τέτοιο, τότε θα πρέπει να θέσουμε ένα αμφιβόλο και το συνολικό πακέτο της μεταρρύθμισης, γιατί για μένα όλα αυτά είναι ένα πακέτο. Μπορούμε να εφαρμόσουμε την αγροτική μεταρρύθμιση υπό την προϋπόθεση και μόνο ότι έχουμε τον απαραίτητο προϋπολογισμό για τα αγροτικά θέματα. Αυτό είναι ένα στοιχείο λοιπόν το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να το θέσουμε στον, ε, στη συζήτηση και είναι κάτι παραπάνω από το καθαρά χρηματικό θέμα. Εγώ σε ευχαριστώ, Πίτερ. Και τώρα ο Αντιπρόεδρος Ζωζέ Μποβέ. Μάλιστα. Πιστεύω πως όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να υπερασπιστούμε έναν σημαντικό γεωργικό προπολογισμό και ότι αυτό ο προπολογισμό θα επιτρέψει την άσκηση πολιτικών. Αν όμω θέλουμε να είμαστε σε θέση να πείσουμε ε, πέρα από τα σύνορα τη επιτροπή μα τα άλλα μέλη αυτού του Κοινοβουλίου, εάν θέλουμε επίση να αντισταθούμε στα κράτη τα οποία θέλουν ενδεχομένω να μειώσουν τον όγκο, θα πρέπει να παρουσιάσουμε, να υποβάλουμε ένα σχέδιο το οποίο να είναι συνεπέ. και γι' αυτό υπάρχουν τρία βασικά στοιχεία των οποίων θα βασιστούμε. Ένα είναι το θέμα τη απασχόληση. Ε, που συνδέεται με το θέμα της κρίσης. Η απασχόληση στον γεωργικό κόσμο θα πρέπει να είναι στην καρδιά του προγράμματός μας. Επίσης, όταν λέμε ότι πρέπει να είναι πιο αγρονομική η γεωργία, να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή και εδώ πάλι πρόκειται για θέμα γεωργικά, για μέτρα γεωργικά και περιβαλλοντικά. Έχω και χρειαζόμαστε κόσμο για να θέσουμε σε εφαρμογή αυτές τις πολιτικές. Και επίσης, ένα τρίτο σημείο, ο υπολογισμό και η οικονομία που μπορούμε να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν είμαστε σε θέση να είμαστε πιο αυτόνομοι για τις, όσον αφορά τι εισαγωγές, θα έχουμε καλύτερο εμπορικό ισοζύγιο. Και αυτό θα πρέπει να μπει στην καρδιά του προγράμματό μα. Ταυτόχρονα, ε, να έχουμε το εμπορικό ισοζύγιο υπόψη μας. Να σας θυμίσω, και θα το έχετε δει μάλλον, στις 19 Σεπτεμβρίου όλες οι ενώσεις που ασχολούνται με τη γεωργία για το περιβάλλον, με το περιβάλλον και με τα ποιοτικά γεωργικά προϊόντα θα είναι εδώ για να συναντήσουν τους ευρωβουλευτές. Είναι απαραίτητο να γίνει αυτή η σύνδεση ανάμεσα στους πολίτες και το κοινοβούλιο μας για να μπορέσουμε καλύτερα να υπερφυστούμε τον ε, προπολογισμό μας. Μάλιστα, ευχαριστώ ε, Ζωζέ Ρόντουστ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρό μας για την πρωτοβουλία που ανέλαβε και να κάνω απόλυτα σαφές ότι δεν είμαι διατεθειμένη να δεχτώ μεγάλες περικοπές στον αγροτικό προϋπολογισμό. Αν θέλουμε το greening, το πρασίνισμα, και θέλω να γίνει κάτι τέτοιο, θέλω να υπάρξει πραγματικό πρασίνισμα της αγροτικής οικονομίας και αυτό κοστίζει χρήματα, άμεσα ή έμεσα. Όταν ζητάω λοιπόν από τους γεωργούς να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα για την, ε, το πρασίνισμα, δεν μπορώ να σου πω συγχρόνως ότι ναι, αλλά θα δεχτείτε και περικοπές στην, ε, στις που παίρνουν. Πρέπει λοιπόν όλοι ενωμένοι να σταθούμε έναντι της Επιτροπής προϋπολογισμού για τα θέματα αυτά. Όταν λοιπόν μας λέει η Επιτροπή ε, Προϋπολογισμών ότι αν υποστηρίξετε το Green το πρασίνισμα, θα είμαστε μαζί μας, μαζί σας και το Συμβούλιο θα είναι μόνος αντίπαλος. Και θα πρέπει να καταλάβει το Συμβούλιο ότι το 30% πρασίνισμα μπορεί να λάβει η χώρα μόνο αν υπάρχει η απαραίτητη χρηματοδότηση. Και αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το θέσουμε σε διαπραγμάτευση. Ο Άλμπερντ Ντες και η Μπρίτα μετά. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για το έγγραφο της νομοδότησης, το οποίο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και εγώ μπορώ να εξάρω αυτά που είπαν προηγουμένως προλαλήσαντε συνάδελφοι από όλε τι πολιτικές ομάδες και έχει δίκιο και ο George Λάιον. αν υπάρξουν ε, περικοπές, αυτές οι περικοπές θα πρέπει να είναι αιτιολογημένε και δεν μπορούν να είναι συλλήβδιν και μόνο στο κεφάλι τη γεωργίας. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε επίση το θέμα τη ξηρασία που σώβει σε μεγάλα μέρη τη Ευρώπη, στην Ουγγαρία, σε τμήμα τη Γερμανία και σε άλλε χώρε. Όλα αυτά δείχνουν πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά και πώς είναι απαραίτητο να ξέρουν οι γεωργοί ότι έχουν κάποια ασφάλεια σε σχέση με τι επιδοτήσει. Γιατί για πολλού απειλείται η ίδια επιβίωσή τους άμα δεν έχουν αυτέ τι επιδοτήσει γιατί μπορεί να βγάζουν 2 τόνους δημητριακά ή 5 τόνους τέφλα. Εάν δεν ξέρουν τι θα προέλθει για τα προϊόντα αυτά, τότε δεν έχουν καμία ασφάλεια σε σχέση με τις επιχειρήσεις τους. Επίσης είναι αδιαμφισβήτητο και το έχουμε δει αυτό μέσα στα πλαίσια της αγροτικής πολιτικής όταν ε, υπάρχει ε, όταν υπάρχει μείωση των επιδοτήσεων και περικοπή προς τους γεωργούς, αυτό οδηγεί σε μια έκρηξη των τιμών και αυτό τελικά αποβαίνει εις βάρος των καταναλωτών στις χώρες μας. Στην Λετωνία την προηγούμενη εβδομάδα είχα πάει να επισκεφθεί ένα συνάδελφό μου και μου έδειξε μια αγροτική εκμετάλλευση που ήταν οικογενειακού χαρακτήρα με 12 αγελάδες και όπου η ιδιοκτήτρια αυτής της φάρμαστον τον ευχαρίστησε για την υποστήριξη που παίρνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και του ζήτησε να βοηθήσει για να έχουν ένα ψυχτικό σύστημα για το γάλα το οποίο παράγουν. Αλλά αυτό το οποίο είναι σαφές από αυτή την, το παράδειγμα που σας δίνω είναι ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε την επιβίωση των γεωργών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να έχουμε μια πολιτική η οποία να μην υφίσταται 30% περισσότερες ε, επιβαρύνσεις για το πρασίνισμα, ενώ συγχρόνως θα πρέπει να αντεπεξέλθει με 20% λιγότερα χρήματα. Δεν μπορεί με αυτόν τον τρόπο να εφαρμοστεί η αγροτική πολιτική από εμά. Ευχαριστούμε. Άλμπερτ Μπρίτα Ρέμερς και μετά η Ελίσσα Σας ευχαριστώ για αυτή την εξαιρετική έκθεση. Τώρα θα ήθελα να προσθέσω ένα στοιχείο μετά από αυτά τα γενικά που ακούστηκαν. Θα πρέπει να πούμε ότι η, η πολιτική γεωργίας έχει επίπτωση στον γεωργικό κόσμο, στην ύπεθρο, στη ε, βιομηχανία. Δεν είναι μόνο ότι πρέπει δηλαδή να στηρίξουμε τη γεωργία, αλλά ότι οι γεωργοί επενδύουν με τρόπο περιφερειακό. Εάν θέλουμε λοιπόν να κερδίσουμε χρήματα, πρέπει να κινητοποιηθεί ο γεωργικός κόσμος. Δηλαδή, δεν είναι πάντοτε τα κορεάτικα τρακτέρα, πιο τοπική παραγωγή θέλουμε να στηρίξουμε. Και εδώ φυσικά είναι ένα επιχείρημα το οποίο πρέπει να ε, επικαλεστούμε. και να δείξουμε και στους συναδέλφους μας πώς η Γεωργία επηρεάζει τους άλλους τομείς. Σε ευχαριστώ. Η Ελίζα Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Και εγώ συμφωνώ με τα όσα είπαν οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ για την πρόταση. Αυτό το σχέδιο ε, έκθεσης, εγώ να πω ότι ε, συμφωνώ μάλλον με την κυρία Ντελάνγκε, ότι δηλαδή πρέπει να κρατήσουμε μια διπλωματική θέση όταν ε, μιλάμε για τα χρήματα για τη Γεωργία. Οι συνάδελφοι είπαν και σωστά ότι το πρασίνισμα, το greening, είναι μια πιθανή λύση μόνο αν δεν υπάρχουν ε, σημαντικές σημειώσεις. Ε, εγώ πιστεύω λοιπόν πως αυτό είναι το προς το συμφέρον μας. Είναι το δικό μας καθήκον να, και αποφύλουμε να ζητήσουμε οι πληρωμές για τους γεωργούς να εξασφαλιστούν για τον καταναλωτή επίσης η γεωργική πολιτική δεν αφορά μόνο τους γεωργούς αλλά και τους καταναλωτές, ολόκληρη την κοινωνία. Και έπειτα κάτι ακόμα που ήθελα να πω ε, για το δεύτερο πυλώνα για την ανάπτυξη της υπαίθρου υπάρχουν πολλές δυνατότητες περικοπών ε, γίνεται λόγος ε, σε όλα τα κράτη-μέλη για αυτά και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τα συζητήσουμε πρέπει να τα συζητήσουμε εν γέννη σε σχέση με τις γεωργικές περιφέρειες. Τα συζητήσαμε και όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της γεωργικής πολιτικής και πρέπει νομίζω να αντιδράσουμε για να διατηρήσει η γεωργία μας. Ευχαριστούμε Ελίζαμπετ. Ο κύριος Μάρτιν Όσλινγκ. Εφόσον ε, εισάγονται περικοπές πλήττεται ο πρώτος πυλώνας. Εμείς πρέπει λοιπόν να αποσαφηνίσουμε στην γνωμοδότησή μας ότι η σημερινή κατανομή θα πρέπει να διατηρηθεί και όσον αφορά το σημείο 7 ε, γίνεται λόγος για ευελιξία. Όμως οφείλουμε να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στον πρώτο και στο δεύτερο πυλώνα ώστε να αποφύγουμε ο δεύτερος πυλώνας να πληγεί περισσότερο. Πρέπει να μην επιτρέψουμε αυτή τη δυνατότητα και αυτό είναι και αυτή είναι και η ουσία της πρότασής μου. Δεν πρέπει να δώσουμε την εντύπωση στα κράτη-μέλη πώς λαμβάνεται μία απόφαση στις Βρυξέλλες και η οποία δεν μπορεί να αλλάξει και δεν μπορούμε να στηρίξουμε ε, αυτές τις περικοπές. Πρέπει να αποσαφηνίσουμε την πρότασή μας. Πρέπει νομίζω να υπάρχει σαφήνεια. Γίνεται λόγος για το πρασίνισμα της γεωργικής πολιτικής και είναι σημαντικός αυτός ο στόχος ε, της μεταρρύθμισης και από αυτό πορέουν, ε, μα εξαρτώνται μάλλον νέες θέσεις απασχόληση. Δεν πρέπει να λέμε πω όλα θα πρέπει να μείνουν όπως είχαν, ότι δηλαδή αφού δεν υπάρχουν χρήματα δεν θα γίνει και καμιά μεταρρύθμιση. Αυτό ω επιχείρημα δεν στέκει είναι αλήθεια πως χρειάζονται επενδύσεις, όμως δεν μπορούμε να πάρουμε πολύ συντηρητική θέση γιατί δεν θα μας βοηθήσει τίποτα. Συμφωνώ μαζί σου Μάρτιν και ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις με τον κύριο Ρούμπιξ. Παρακαλώ un finanšu sadalījumu 2014. gadā. Θα ήθελα να μιλήσω για το θέμα της κατανομής των χρημάτων ε, για την περίοδο 2014 με 2020. Το ξέρουμε πάντα εδώ και πολύ καιρό ότι είναι έτσι και πάντα θεωρήσαμε ότι πρέπει να υπάρξει μεταρρύθμιση στην κοινή αγροτική πολιτική και αυτό είναι κάτι το οποίο προσδοκούν και οι ίδιοι οι γεωργοί. Εγώ έχω επισκεφθεί πολλούς γεωργούς στη Λετωνία πρόσφατα, πρόσφατα και υπάρχουν πολλές προσδοκίες. Αυτά που είπε ο κύριος Ντες είναι απόλυτα έγκυρα. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο βλέπει κανείς όταν συναντάει τους γεωργούς. Περιμένουν όλοι ότι θα γίνει κάτι και ότι θα πραγματοποιηθεί η μεταρρύθμιση. Αλλά όπως έχουν αυτή τη στιγμή τα πράγματα, αυτή η μεταρρύθμιση θα τους πλήξει ιδιαίτερα σκληρά. Εγώ θα ήθελα να βρούμε ένα πιο διπλωματικό τρόπο να εκφράσουμε την απόψή μας στο έγγραφο αυτό, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι σε σχέση με τους στόχους που επιθυμούμε να επιτευχθούν. Αν περικόψουμε τα κονδύλια στην Γεωργία, θα φέρουμε και την ευθύνη για τις περικοπές αυτές ή τουλάχιστον θα φανούμε σαν να είμαστε εμείς οι υπεύθυνοι για αυτές τις περικοπές. Γι' αυτό εγώ θέλω να τονίσω την απόλυτη αντίθεσή μου από τη μία πλευρά να περικόπτονται τα κονδύλια στη γεωργία ενώ συγχρόνως σπαταλώνται απόλυτα τεράστια ποσά για στρατιωτική έρευνα ή στρατιωτική πολιτική. Συμφωνώ λοιπόν και με τους προλαλήσαντες συναδέλφους και φυσικά υποστηρίζω τη θέση του Πρόεδρου. Σας ευχαριστούμε κύριε Ρούμπιξ. Ο Λουίς Καπούλα Σάντος για να κλείσει. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι δύσκολο να προσθέσει κανείς κάτι ακόμα στα όσα είπαν ήδη οι συνάδελφοι. Θα ήθελα να υπογραμμίσω την μεγάλη συνένεση ε, που επικρατεί για αυτή την έκθεση και να την ε, ενισχύσουμε μάλιστα τη θέση αυτή. Επανειλημμένως έχουμε κρατήσει εξάλλου αυτή την ε, θέση και ελπίζω αυτή η συνένεση σε αυτό το θέμα να παραμείνει και να διευρυνθεί για τα βασικά θέματα επί των οποίων θα χρειαστεί να αποφασίσουμε σε λίγο όσον αφορά το μέλλον της γεωργίας και των Ευρωπαίων γεωργών. Νομίζω πως ε, η συγγήτρια σωστά ερμήνευσε την ε, βούληση όλης της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ. Τώρα θα δώσω το λόγο στον ε, Διευθυντή Λόγκο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να σχολιάσω την έκθεση την οποία ετοιμάσατε, την οποία διαβάσαμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λάβαμε πολύ προσεκτικά διάφορα συμφέροντα τα οποία τα εξετάσαμε πολύ αναλυτικά. Ακούσαμε και σήμερα τις αντιδράσεις σας στη συζήτηση, τις οποίες θεωρούμε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και φυσικά θα τις ε, αναφέρω και στους ανωτέρους μου. για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τα όσα λέγονται είναι πολύ σημαντικά για την κοινή γεωργική πολιτική, διότι προφανώς ε, αποτελούν τη βάση της και επιτρέπουν ε, να διασφαλίσουμε το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής υπό τους άρους μιας ισχυρής κοινή γεωργικής πολιτικής. Επομένως, η χρηματοδοτική πρικοδότηση είναι ιδιαίτερα σημαντική. Θα ήθελα να υπενθυμίσω δύο σημεία ε, τεχνικής ε, σημασίας απλώς και μόνον που αφορούν την έκθεση. Να σας πω απλώς ότι για το 2007-2013 ο καθορισμός για το ταμείο είχε καθοριστεί το 2002. Η ε, συνεισφορές που είχαν αποφασιστεί είχαν ε, καθορίσει ότι για την κυνηγή η γεωργική πολιτική θα υπήρχε μείωση σε πραγματικούς όρους διότι η προσαρμογή για τον αποπληθωρισμό δεν ήταν ε, ε, πραγματική αλλά ήταν μερική. Επομένως πρέπει να λάβουμε υπόψη και αυτή την πτυχή αν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε σύγκριση μεταξύ του 2007 και του 2013 και του 2014-2020. Επιπλέον, θα ήθελα να διευκρινίσω, απαντώντας σε κάποιες από τις παρατηρήσεις που έγιναν, ότι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2014-2020 παρουσιάστηκαν ευθύς εξ αρχής ως πάγωμα αλλά σε σχέση μόνο με το 2013 και όχι για το σύνολο της περίοδου. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω ότι οι απαραίτητες ε, συνεισφορές ε, οι οποίες πρέπει να γίνουν λόγω της ένταξης της Κροατίας έχουν ε, ληφθεί υπόψη στην επικαιροποίηση της πρότασης προϋπολογισμού για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο την οποία ενέκρινε προσφάτως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω στις 6 Ιουλίου αν δεν κάνω λάθος. Θα ήθελα λοιπόν να περιοριστώ σε αυτά τα στοιχεία, τα οποία είναι απλώς στοιχεία και θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς και τους συναδέλφους σας κύριε Πρόεδρε για την ε, γνωμοδότηση και για την πολύ ενδιαφέρουσα, επαναλαμβάνω, σημερινή συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Διευθυντή Λόγκο και θα λάβουμε υπόψη του και τις διευκρινήσεις που μας έκανε. Να σας υπενθυμίσω για άλλη μια φορά ότι αύριο στις 12 λίγη η προθεσμία κατάθεσης ε, τροπολογιών. 4 Σεπτεμβρίου, 12 το μεσημέρι. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι και ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους που έλαβαν το λόγο. Να επανέλθουμε τώρα στο σημείο 4 της ημερίας διάταξης, όπου ζητώ συγγνώμη από τη συνάδελφο Λάγκε, αλλά επειδή έπρεπε να ε, ψηφίσουμε, ξέχασα ότι πρέπει να κάνουμε και συζήτηση για το σχέδιο της νομοδότησης το οποίο θα ψηφίσουμε ε, στις 18 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στην κυρία Ντελάνγκη για να μας παρουσιάσει απόψεις της. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επειδή η ψηφοφορία για τις γραμμές ε, του προπολογισμού ε, πήγε ακριβώς βάσει των όσων είχαμε συζητήσει μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Το σχέδιο της γνωμοδότησης δεν χρειάζεται να τροποποιηθεί πάρα πολύ αναλυτικά, διότι δεν έχουμε πολύ ψηφίσει και πολλά πράγματα αντίθετα στο σχέδιο γνωμοδότησης. Βέβαια δεν πάβει να υπάρχει η προθεσμία για την κατάσταση των τροπολογιών, η αυριανή προθεσμία ε, και ίσως ε, να υπάρχουν κάποια θέματα στα οποία θα ήθελαν να αναφερθούν οι συνάδελφοι μέσω τροπολογιών τους. Αυτό που κάνει αυτή η γνωμοδότηση είναι να διευκρινίζει ότι η γεωργική πολιτική δεν είναι η μεγαλύτερη αύξηση για το 2013. Γίνεται μεγάλη συζήτηση για τη συνολική αύξηση κατά 7% των πληρωμών. Άμα δείτε ε, για τον πρώτο πυλώνα της γεωργικής πολιτικής έχουμε 0,5% και ένα 2% είχαμε για την ανάπτυξη υπαίθρου. Επειδή όμως είναι πολύ σημαντική η συζήτηση επί του προπολογισμού που γίνεται ε, αυτή τη στιγμή, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Και αυτό κάναμε με αυτή την ψηφοφορία. Δεν υπερψηφίσαμε μόνο κάποιες προτεραιότητες που θεωρούμε εμείς ότι είναι πολύ σημαντικές για την Επιτροπή μας, αλλά ψηφίσαμε και μείωση κάποιων ε, γραμμών προπολογισμού. Έχουμε λοιπόν δείξει ότι μπορούμε να περιοριστούμε, έχουμε ε, καθορίσει κάποια κονδύλια για τις ε, επιστροφές, για τις αποζημιώσεις, ε, για να μπορούμε να έχουμε επιπλέον πληρωμές και θα ήθελα αυτό να το σημειώσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα τονίσουμε και κάτι τέτοιο και στην Επιτροπή Προπολογισμών και στο Συμβούλιο. Για παράδειγμα, στον τομέα των φρούτων και των απορροκυπευτικών όπου υπήρχαν αντίξωες συνθήκες, υπήρχαν αντιδράσεις και από την Ισπανία και από την Ανατολική Ευρώπη, κάτι πρέπει να γίνει από αυτόν. Εάν έχουμε ε, ε, μια απολευθερωμένη κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει ε, να διαβιβάζεται ε, το μήνυμα αυτό περισσότερο στους ανθρώπους που αγοράζουν τα προϊόντα. Οι καταναλωτές λοιπόν πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλύτερα τι συμβαίνει και αυτό θα πρέπει να το κοινοποιήσουμε στην Επιτροπή Προπολογισμών. Στην γνωμοδότηση ε, διευκρινίσαμε και το συζήτησα επανειλημμένως και μαζί σας αυτό θεωρούμε ότι τα πιλωτικά προγράμματα τα οποία υπερψήφισε το Κοινοβούλιο θα πρέπει να υλοποιηθούν. Ε, γίνονται και κάποιες προτάσεις για το πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και ποια είναι τόσο πολύ σημαντικά για μας ως Επιτροπή Γεωργίας. Ε, επιπλέον να σας πω ότι ε, νεκρήθη ένα επιπλέον πιλωτικό πρόγραμμα από πλευράς Πρασίνων για τις ε, ε, γενετικούς πόρους και προτείνω να ληφθεί υπόψη και αυτό ε, στην ψηφοφορία μας. Με αυτό λοιπόν ολοκληρώνω την παρέμβασή μου και προσβλέπω στα σχόλια των συναδέλφων. Ευχαριστώ Έστερ. Με τη διευκρίνηση αυτή λοιπόν για το σχέδιο γνωμοδότησης, εάν δεν υπάρχουν ε, κάποιες άλλες παρεμβάσεις ε, και δεν υπάρχει κάποιος άλλος που να θέλει να λάβει το λόγο, μπορούμε να επανέλθουμε στη συνέχεια της μερίσιας διάταξης, εκεί που διακόψαμε και πάμε στο σημείο 7. Περνάμε στο ψωμί λοιπόν. Άμεσε πληρωμέ υπέρ των γεωργών στο πλαίσιο των καθεστώτων στήριξη τη κοινή γεωργική πολιτική. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπω γνωρίζετε, πριν από τι θερινέ διακοπέ, ε, είχαν γίνει κάποιε εκτιμήσει. Είμαστε ήδη άνω των 7.000 τροπολογιών πλέον, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που παρουσίασαν οι εισηγητές. Ε, Αυτές λοιπόν είναι όλες οι τροπολογίες που έχουμε συλλέξει για τις τέσσερις βασικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό καταδεικνύει βέβαια πόσο σημαντική είναι η μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής και πόσο είμαστε όλοι μας διατεθειμένοι να βελτιώσουμε το κείμενο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνοντας βεβαίως υπόψη και τις ποικιλομορφίε της γεωργικής πολιτικής ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημαντικό λοιπόν είναι να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς που θα μας οδηγήσουν σε ισορροπημένες λύσεις για όλο το γεωργικό τομέα και θα μπορέσουμε να δώσουμε μια ενωμένη στεναρή εικόνα ως Ευρωπαϊκό Βούλιο για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που είχαμε κάνει και στο παρελθόν με τις εκθέσεις του George Lyon και του Albert Dess. Δεν θα είναι βέβαια πανεύκολο μόνο για το θέμα αυτό, για τις άμεσες ενισχύσεις, έχουμε 2.292 τροπολογίες, εκ των οποίων 111 τροπολογίες είναι του Λουίς Μανουέλ Καπούλα Σάντος, τον οποίο θα δώσω το λόγο εντός ολίγο, και 500 τροπολογίες αφορούν το greening, το μετριασμό των, συνθηκών, των επιπτώσεων του περιβάλλοντος στη Γεωργία. Θέλουμε λοιπόν να ε, καταλήξουμε σε συμβιβασμούς και να δώσουμε την εικόνα μιας ενωμένης επιτροπής, αυτό που ελπίζω ότι δώσαμε ως μήνυμα και μέχρι σήμερα. Ελπίζω να έχει έρθει εδώ ο Διευθυντής ο κύριος Πατσέκο και να δώσουμε απευθεία το λόγο στο Λουίς για να ξεκινήσει η συζήτηση. Να σας υπενθυμίσω πριν δώσω το λόγο στο Λουίς ότι αν έχουμε αρκετό χρόνο και αν καταφέρουμε να περιορίσουμε τη συζήτηση για το σημείο αυτό στη μία ώρα περίπου, μία με μία μισή ώρα, θα ήθελα να εξοικονομήσουμε λίγο χρόνο για να κάνουμε μια διευρυμένη ε, συνεδρίαση των συντονιστών με τους εισηγητές για να συζητήσουμε τη στρατηγική διαχείριση αυτών των περίπου 7.000 τροπολογιών. Ευχαριστώ πολύ. Λουίς, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ελπίζω ότι όλοι είχατε ευχάριστες ε, διακοπές και ερχόσαστε με φορτισμένες τις μπαταρίες σας γιατί θα χρειαστούμε πάρα πολύ ενεργητικότητα και προσπάθεια τις επόμενες εβδομάδες για να μπορέσουμε να φέρουμε σε αίσιο πέρα στη συνεργασία μας. Βέβαια σήμερα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να συζητήσουμε το περιεχόμενο των τροπολογιών. Ξέρω ότι δεν είχατε την ευκαιρία να δείτε αναλυτικά όλες αυτές τις ε, τροπολογίες, τον τεράστιο αυτό αριθμό τροπολογιών. Δεν είναι ακόμα διαθέσιμες όλες οι τροπολογίες σε όλες τις ε, επίσημες γλώσσες. Αλλά, εν πάση νομίζω ότι έχοντας αναγνώσει μερικές εκατοντάδες προτάσεων, βλέπει κανείς ότι υπάρχουν ουσιαστικές προτάσεις τροποποίησης, τυπικού χαρακτήρα προτάσεις τροποποίησης, αλλά και προτάσεις οι οποίες εκφεύγουν τελείως από τη λογική μέσα στην οποία εργαζόμαστε για το μέλλον της κοινή αγροτικής πολιτικής. Εγώ θα πίστευα λοιπόν κύριε Πρόεδρε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη σημερινή συνεδρίαση να καθορίσουμε ορισμένες οδικές γραμμές για την εργασία μας, ξεκινώντας από την βασική αρχή, ότι όπως θέλαμε και να το κάνουμε, καταρχήν να ψηφίσουμε σε μία από τις δύο συνεδριάσεις μας του Νοεμβρίου, 5 και 26 Νοεμβρίου, και από ό,τι καταλαβαίνω η πρόθεσή μας είναι τότε το Νοέμβριο να ψηφιστούν οι εκθέσεις αυτές. Επομένως έχουμε στη διάθεσή μας το Σεπτέμβριο αλλά και τον Οκτώβριο που θα απαιτήσουν μια πάρα πολύ έντονη εργασία, πάρα πολύ έντονες διαπραγματεύσεις και αυτό το οποίο θα ήθελα να προτείνω είναι να ξεκινήσουμε το ταχύτερο δυνατό από την επόμενη εβδομάδα να συναντήσω όλους τους ε, σκιώδεις εισηγητές και μετά να περάσω σε διμερείς επαφές με τους ε, σκιώδεις εισηγητές από κάθε πολιτική ομάδα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν να εξετάσουμε όλες τις τροπολογίες, τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε κοινέ θέσεις για τα σημαντικότερα θέματα, όταν υπάρχουν διαφορές οι οποίες μπορούν να γεφυρωθούν με συμβιβαστικές ε, προτάσεις, αλλιώς θα πρέπει να δώσουμε στην Επιτροπή εναλλακτικέ θέσεις για την ψηφοφορία. Εγώ φυσικά είμαι απόλυτα στη διάθεση όλων για να επομιστώ το έργο αυτό και να ανταποκριθώ στις προτάσεις όλων εφόσον δεν, τεθ, δεν θέτουν ένα αφιβόλω τη συνεκτικότητα της έκθεσης. γιατί θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συγκεράσουμε όλες τις απόψεις και τα συμφέροντα τα οποία βρίσκονται επιτάπτως αυτή τη στιγμή και έχουμε ένα τιτάνιο έργο. Φυσικά, όπως είπε και ο πρόεδρος, ανέφερα ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε 7.000 ε, τροπολογίες συνολικά και αυτό σημαίνει μια τεράστια προσπάθεια από την πλευρά όρων μας. Εγώ σας λέω ότι ήδη αυτή τη βδομάδα θα προσπαθήσω να καθορίσω τις ημερομηνίε συνάντησης με τους σκιώδεις εισηγητές και σας κάνω μια έκκληση να προσπαθήσετε να βρείτε τις κατάλληλες στιγμές στο χρονοδιάγραμμά σας, στην ατζέντα σας, ώστε να συναντηθούμε σε αυτές τις ημερομηνίε, γιατί το έργο των σκιωδών εισηγητών θα πρέπει να προχωρήσει κατά προτεραιότητα. Εγώ έχω ακυρώσει όλες τις ε, άλλες μου υποχρεώσεις μέσα στο επόμενο δίμηνο, γιατί είναι σαφές ότι πρέπει εάν θέλουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα, να εργαστούμε σκληρά για την πολιτική διαπραγματεύση αυτό το θέμα. Ωραία, Λουίς, όντω ε, θα είναι μια πολύ περίπλοκη δουλειά, αλλά ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε το τρόπο να αποδείξουμε πως το Κοινοβούλιο έχει μια ξεκάθαρη δική του φωνή και δεν ε, χωρίς αντιφάσει. Θα ξεκινήσω λοιπόν με τους κοιόδες εισηγητές. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Μαγκίνες, την οποία χαιρετώ, και μετά τον Τζόρτζο Λάιον. Συμφωνείτε? Ωραία. Μάριαν, ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εισηγητή μας. Καταρχήν να πω ότι είναι πολύ βοηθητικό το ότι είναι ανοιχτό στις ε, προτάσεις και είπατε ότι είναι πολύ το πολύ περίπλοκο στη γλώσσα σας και όντως είναι. Ε, όμως μπορούμε να απλοποιήσουμε πολύ μεγάλο κομμάτι της δουλειάς μας γιατί έχω δει τις ε, τροπολογίες και έχω δει ότι υπάρχουν ε, επικαλύψεις πολλές. Αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό και ο συγητής το ανέφερε, αυτό είναι η μέθοδος που θα ακολουθήσουμε. Για να έχει νόημα για τους συναδέλφους πρέπει να μπλοκάρουμε κάτι από το κάθε άρθρο της τροπολογίας. Και αυτό είναι δύσκολη δουλειά για την ε, γραμματεία, αλλά αν το καταφέρουμε μπορούμε να λάβουμε τις κατάλληλες πολιτικές αποφάσεις. Αλλά νομίζω πως είναι απαραίτητο να προοδεύσουμε, να προχωρήσουμε. Αν δει κανεί τα επίμαχα ζητήματα, ε, το πρασίνισμα με 600 τροπολογίες, μόνο αυτό, φαντάζεστε ότι θα πρέπει να χρειάζεται πολύ χρόνο να ασχοληθούμε με αυτό, Υπάρχουν ε, εκατοντάδες για πολύ μικρά θέματα, για κάποιες παραγράφους, αλλά πολύ σημαντικές παραγράφους. Άρα λοιπόν πιστεύω πως αυτό η μέθοδος εργασίας θα είναι θέμα κλειδί. Πρέπει πρώτα γι' αυτό να αποφασίσουμε. Θα πρέπει επίσης από πολιτικής άποψης να εκφράσουμε την ανησυχία μας για τα κυπριακά συμπεράσματα την περασμένη εβδομάδα ε, για τον προπολογισμό. Ε, την πρόταση ότι είναι αναπόφευκτες οι περικοπές στον ε, προπολογισμό της Γεωργίας για να παραθέσω τα όσα είπαν οι Κύπροι διαπραγματευτές και περικοπές στις άμεσες πληρωμές και στις, ε, στον πυλώνα της ανάπτυξη πέθρου. Αν λοιπόν βασιστούμε σε αυτό το υπόβαθρο δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα ούτε στο πρασίνισμα ούτε στη σύγκληση ούτε σε τίποτα εάν τελικά περάσει. Η Επιτροπή μας λοιπόν θα πρέπει να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τις απόψεις μας όσον αφορά την κατάσταση του προπολογισμού. Πολύ δύσκολη η κατάσταση ήταν φέτος ε, για τους γεωργούς σε πολλά μέρη της ε, Ευρώπης. Πρέπει λοιπόν να, να στηρίξουμε τη δουλειά μας ε, στις ενδείξεις ε, κατεύθυνσης της συζήτησης περί περιπολογισμού ε, Για να συνοψίσω λοιπόν θα ήθελα να πω πέρα από τα σχόλια όσον αφορά το έγγραφο εργασία να πω ότι γνωριζόμαστε αρκετά καλά ε, μεταξύ μας εδώ στην Επιτροπή όσοι διαπραγματευόμαστε και γι' αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε κάποιες από τις πιο ξεκάθαρες ε, πτυχές ώστε να μπορούμε να συμφωνήσουμε είτε σε διμερείς ε, εδώ αρχίζω και τραγουδάω κανονικά με αυτή τη μουσική, λέει η κυρία Μαγκίνες και θα υπάρξει και ταξιδάκι στη Νέα Υόρκη ε, για όποιους ε, κερδίσουν στην κλήρωση. Λοιπόν, μάλλον θα χρειαστεί να είμαστε έτσι κάπως πιο χαλαροί και να χρησιμοποιήσουμε την αίσθηση του χιούμορ μας για να τα βγάλουμε πέρα εδώ πέρα. Ε, θα πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε με τη μέθοδο και μετά όσο όταν θα περάσουμε στα πιο επίμαχα ζητήματα να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πιο πολύ. Τελευταίο μου σχόλιο είναι ότι το Κοινοβούλιο ψήφισε με συγκεκριμένη κατεύθυνση για το τομεί κλειδιά και πρέπει να αποφασίσουμε αν πρέπει να μείνουμε σε αυτέ τι γραμμέ. Για παράδειγμα, ένα μενού πρασινίσματο. Ξέρω ότι με, για διάφορους λόγους, πολλούς και διάφορους λόγους με, απομακρυνθήκαμε από αυτό. Τώρα αλλάζουμε τελικά την κατεύθυνσή μας ή όχι. Οι δικές μου τροπολογίες έχουν επιμείνει στην ε, ψήφο του Κοινοβουλίου για το θέμα. Ε, θα ήταν λοιπόν καλό να ξεκαθαρίσουμε την θέση του Κοινοβουλίου. Ποια ήταν η θέση μας μέχρι τώρα και αν θα προχωρήσουμε προς αυτή την ατζέντα ή αν θα απομακρυνθούμε. Και επίσης να έχουμε και το, την κατάλληλη εντολή για να το κάνουμε αυτό. Ναι, είναι τεράστιο το έργο, αλλά δεν είναι και ξεπέραστο. Οι βασικές μου ανησυχίες αφορούν τον προϋπολογισμό. Και σίγουρα μπορούμε να περιμένουμε, δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους γεωργούς να κάνουν περισσότερα με λιγότερα χρήματα. Ο εισηγητή έχει, έχει δείξει την προθυμία του να συνεργαστεί μαζί μας πριν από την έκθεση και κατά τη διάρκεια της εκπόνηση της έκθεσή του. Ε, θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τη μέθοδο και το χρονοδιάγραμμα να συμφωνήσουμε για αυτά και μετά στη... θα έχουμε κάθε ομάδα τα δικά της ε, θέματα και τις κόκκινες γραμμές της αλλά θα πρέπει μάλλον να τα συζητήσουμε σε επόμενη συνεδρίαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Μάρεντε, ούτε ή άλλω, ε, πριν από λίγο τα συζητήσαμε αυτά όταν ε, παρουσιάσαμε το σχέδιο γνωμοδότησης ε, για, και για τον Ε, πρόκειται για πρόταση που περιλαμβάνει περικοπές, όχι για πάγωμα. Εάν υπάρξουν τόσο σημαντικές λοιπόν περικοπές και εγώ αμφιβάλλω ε, τι θα γίνει με τη μεταρρύθμιση και το πρασίνισμα. Ο George Λάιον και μετά ο κύριος Όσλινγκ. Uh, thank uh, uh, Σας ευχαριστώ και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τις προτάσεις του σε σχέση με τη συνεργασία των σχεδόν εισηγητών και τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουμε να πετύχουμε μεγαλύτερη πρόοδο στο θέμα αυτό από τη δική μας οπτική γωνία ως Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν έχουμε 7,5 ή 8.000 ίσως τροπολογίες πια. Το βασικό θέμα είναι να μπορέσουμε στο τέλος να βγάλουμε κάτι από, αυτή την, από αυτό το κείμενο που δεν είναι μια γνωμοδότηση, είναι ένα νομικό κείμενο, το οποίο όμως ε, να έχει μια συνεκτικότητα, γιατί αυτό θα καθορίσει τη ζωή των γεωργών μας τα επόμενα 7 χρόνια και θα παίξει και ένα σημαντικό ρόλο για την εξέλιξη της κοινή αγροτικής πολιτικής μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τεράστια η ευθύνη λοιπόν που έχει αναλάβει το Κοινοβούλιο μας ώστε να εξασφαλίσει ότι θα βγει ένα αξιόπιστο και συνεκτικό κείμενο από αυτή την προσπάθεια και να είναι κάτι το οποίο μπορούν πράγματι να εφαρμόσουν οι γεωργοί μας. Είναι λοιπόν μια τεράστια πρόκληση, όπως λέω, να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι συνεκτικό και αξιόπιστο αυτό το έγγραφο το οποίο θα προέλθει από την ψηφοφορία. Δεν μας βοηθάνε οι 7.500 τροπολογίες προφανώς. Και εδώ χρειάζεται η σωστή μεθοδολογία και νομίζω ότι αυτά που πρότεινε ο εισηγητής μας βοηθούν. Αν δείτε τις τροπολογίες, βλέπω το άρθρο 4, αλλά έχει 25 σελίδες τροπολογίες για ουσιαστικά τον ίδιο τομέα. Για τέτοιες τροπολογίες που είναι τεχνικές και όχι πολιτικής σημασίας μπορούμε να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα εφόσον έχουμε μια σαφή εικόνα του τι θέλει ο καθένας που καταθέτει τροπολογία. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε πρόοδο για τα θέματα αυτά και να αφήσουμε τα πραγματικά πολιτικά επίμαχα θέματα προς το τέλος. Και χρειαζόμαστε ειδικό χρόνο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις τροπολογίες. Και φυσικά το ερώτημα είναι αν θα ακολουθήσουμε την πολιτική γραμμή που έχουν δείξει οι προηγούμενες εκθέσεις ή αν θα έχουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση χάρη για το θέμα της ε, προστασίας του περιβάλλοντος, το greening. Η ομάδα μου λοιπόν υποστηρίζει το να εργαστούμε ως το δυνατόν πιο σκληρά για να καταλήξουμε σε συμβαστικές λύσεις, ώστε να μπορούμε στη συνέχεια να περάσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες εγκαίρως, ώστε να είμαστε έτοιμοι για τις διαπραγματεύσεις πρώτης ανάγνωσης. Αν το Συμβούλιο θέλει να ξεκινήσει τα Χριστούγεννα, εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι με το τελικό μας κείμενο τα Χριστούγεννα. Αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή μας θα πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις πριν από το τέλος του έτους. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Εγώ είμαι πρόθυμος να εργαστώ όσο σκληρά απαιτείται για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Σίγουρα. Έχει χρειαστεί τόσο πολύ καιρό για να προχωρήσουμε προς την μεταρρύθμιση αυτή που σίγουρα πρέπει να φέρουμε αυτή την ε, προσπάθεια σε ένα αίσιο πέρας. Αυτό εν μέρη δικαιολογεί και αυτή την πλημμυρίδα τροπολογιών. Είναι πολύ σημαντικό για το Κοινοβούλιο λοιπόν να παίξει ένα σημαντικό ρόλο, ακόμα και αν αυτό μας φέρει αντιμετωπούς σε μια τεράστια πολυπληθώρα τροπολογιών, σε μια απόλυτη πληθώρα απόψεων. Πιστεύω όμως ότι αυτό θα πρέπει να γίνει και με μια εσωτερική, κατά κάποιο τρόπο, προετοιμασία μέσα στις πολιτικές ομάδες, ώστε οι σκιώδεις συζητητές να μπορούν να μεταφέρουν τις απόψεις των δικών τους βουλευτών. Το χρονοδιάγραμμα που έχουμε ενώπιόν μας δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Γι' αυτό θα πρέπει να ξεχωρίσουμε την ήρα από το στάρι, να αφήσουμε τα θέματα τα οποία είναι τεχνικά από τα θέματα που είναι πολιτικά, να δώσουμε την έμφαση στα θέματα του greening, όλα αυτά τα ζητήματα που βρίσκονται και στον πρώτο πυλώντα. Και το βασικό θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι φυσικά αυτό της μεταρρύθμισης. Τα θέματα του προπολογισμού είναι χωριστά, αλλά όπως είπε και η κυρία Μαγκίνες, δεν μπορούμε να αποσυνδέσουμε το ένα από το άλλο. Δεν μπορεί να γίνει μεταρρύθμιση χωρίς χρηματοδότηση. Δεν μπορούμε να απλοποιήσουμε τα πράγματα σε τέτοιο σημείο. Πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να προωθήσουμε τα θέματα της μεταρρύθμισης, ενδεχομένως με λιγότερα κονδύλια στη διάθεσή μας. Υπάρχει ένα άλλο σημείο, το οποίο είναι η αίτηση των συναδέλφων από, την, από τα νέα κρατημέλη που ζητούν να προασπιστούν τα κονδύλια τα οποία δίνονται προς τις χώρες τους, κάτι που είναι απαραίτητο. Αν μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό ή όχι, αυτό δεν είναι δεδομένο. Πιστεύω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς ώστε να μην αφαιρέσουμε όλα τα ποσά από τους υπόλοιπους, ενώ συγχρόνως λέμε και στα νέα κράτη ότι δεν μπορούμε να καλύψουμε όλες τις απαιτήσει τους. Τις επόμενες εβδομάδες θα πρέπει οι πολιτικές ομάδες να δούνε ποια είναι τα κύρια σημεία, τα κέρια σημεία στην πρόταση αυτή. Για ορισμένου είναι το να υπάρξει μια εξοικονομήση κονδυλίων. Παραδείγματος χάρη. Και να αφήσουμε όλα τα θέματα τα οποία είναι τα πιο επίμαχα για να μείνουν στο τέλος. Είναι απαραίτητο όμως εμείς να πάρουμε την, την τελική απόφαση εγκαίρως. Γιατί αλλιώς το Κοινοβούλιο θα χάσει την αξιοπιστία του. Αν δεν μπορέσουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα, δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα καθυστερήσει παραγωγικά το Συμβούλιο και ότι θα έχουμε αρκετό χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο. Θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι πρέπει να κλείσουμε την εργασία μας το ταχύτερο δυνατό. Ευχαριστώ Μάρτιν, η Έστερ και στη συνέχεια οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι αφιερώνουμε αυτή τη συνεδρίαση για να συζητήσουμε πώς θα συζητήσουμε τα πράγματα. Διότι ουσιαστικά αυτό κάνουμε. Και έχουμε καθυστερήσει, έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ σε σχέση με τις υπόλοιπες επιτροπές. Και εάν δεν βιαστούμε θα βρεθούμε εκτός συζήτησης και όχι εντός συζήτησης. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέει ο Μάρτιν Χάουσλινγκ ότι οι πράσινοι συμφωνούν μεταξύ των, αλλά αυτό δεν σου δίνει τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργική πολιτική. Μια ομάδα μόνη τη δεν αποφασίζει. Έχω να κάνω μια πρόταση λοιπόν. Νομίζω ότι ήταν πολύ σαφή τα πράγματα στα θέματα της αλληλοεπικάλυψης και της κατάλληλης διάρθρωσης και από τον ε, εισηγητή για το θέμα αυτό ακούω ότι θέλει να συζητήσει με τους κοιόδης εισηγητές. Αυτό είναι λογικό. Αλλά πριν συζητήσει με αυτούς θα πρέπει να υπάρχει μια σαφής δομή η οποία θα παρουσιαστεί σε όλα τα μέλη ώστε να γνωρίζουμε γιατί ακριβώς συζητάμε. αυτό που κάνουμε στην, ε, στο κόμμα μου, όταν γίνεται συνέδριο του κόμματος, είναι ότι έχουμε ε, κάποιες ε, τροπολογίες οι οποίες είναι πρώτη κατηγορίες και η γραμματεία θα μπορούσε απλώς να τις ε, ε, περάσει αμέσως και υπάρχουν οι δεύτερες μορφής τροπολογίες οι οποίες απαιτούν περισσότερη συζήτηση. Τα βασικά συζητήματα όμως είναι τροπολογίες τρίτου τύπου και πάλι όμως εκεί η γραμματεία θα μπορούσε να διευκρινίσει ποια είναι τα διάφορα φιλοσοφικά ρεύματα. Για παράδειγμα, για το greening ποιες είναι οι τάσεις και από εκεί και πέρα να δούμε τα υπόλοιπα. Και έτσι θα μπορούν οι εισηγητέ και οι σκιώδει εισηγητέ να συζητούσουν μεταξύ του. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια διαφάνεια, διότι νομίζω ότι επικρατεί διαφάνεια εδώ. Δεν μπορούμε να παρουσιάσουμε μια διαπραγμάταξη μεταξύ 5-6 ατόμων πρώτα στην Επιτροπή και μετά στο Κοινοβούλιο και να του πούμε ή υπερψηφίστε την ή καταψηφίστε την. Θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλου και εδώ στην Επιτροπή αλλά και ευρύτερα στο Κοινοβούλιο να γνωρίζουν τι ακριβώ συζητούμε, πού επικεντρωνόμαστε και θα πρέπει να υπάρχει μια σαφή εικόνα και μια δομή για να ξέρουμε γιατί ακριβώ συζητάμε. Και νομίζω, κύριε Πρόεδρε, ε, και λυπάμαι που το λέω την πρώτη μέρα των συνεδριάσεων μετά το θερινό διάλειμμα, χρειαζόμαστε και άλλε συνεδριάσει. Πρέπει να παρατήσουμε αυτά που κάνουμε για να συναντιόμαστε συχνότερα, ιδίω για αυτά τα τρίτη κατηγορία θέματα που είναι τα πιο διαφιλονικούμενα. Ευχαριστώ, Έστερ, αλλά αυτή την πρόταση έκανα και προηγουμένω. Αν καταφέρουμε να τελειώσουμε τη συνεδρίαση τη Επιτροπή μα αρκετά νωρί, θα ήθελα να συζητήσω με του συντονιστέ και του ε, εισηγητέ μια μέθοδο και από εκεί και πέρα να οργανωθούμε ε, με την ουσιαστική συνεισφορά της ε, γραμματείας που θα πρέπει να μας βοηθήσει να διαρθρώσουμε και να έχουμε ένα σύστημα για όλες αυτές τις τροπολογίες, πολλές από τις οποίες είναι διπλές ή και τριπλές. Ähm, Εγώ βλέπω ότι εδώ είμαστε έτοιμοι να φάμε όλοι μας το χρόνο για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό στο Κοινοβούλιο, τι θα κάνουμε με τον προϋπολογισμό, αλλά περί της μεταρρυθμίσεως λόγος ουδής. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν και υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία είναι επίμαχα όχι μονάχα μεταξύ των πολιτικών ομάδων αλλά και μέσα στις ίδιες τις πολιτικές ομάδες. Δεν θα πρέπει λοιπόν παρά τις ιδιαίτερες πιέσεις τις χρονικές που έχουμε ενώπιόν μας να ξεχάσουμε αυτά τα σημεία. Θα πρέπει να σκεφτούμε πόσο πρακτικά και εφαρμόσιμα θα είναι τα μέτρα αυτά τα οποία πρέπει να εφαρμόσει ο Γεωργός. Δεν αρκεί να είμαστε σωστοί εναντί του Κοινοβουλίου και να καλυφθούμε μέσα στα πλαίσια του προπολογισμού και να μην ξεχάσουμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια τεράστια γραφειοκρατία η οποία ουσιαστικά ταλανίζει τους γεωργούς και δημιουργεί πρόσθετο κόστος. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για τη μείωση της γραφειοκρατίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί αυτό θα οδηγήσει και σε μεγαλύτερη αποδοχή από την πλευρά των γεωργών και γενικά των Ευρωπαίων πολιτών. Θέλουμε λοιπόν να κάνουμε κάτι το οποίο θα βοηθήσει την Ήπεθρο ή θέλουμε απλώς να έχουμε μια γραφειοκρατία η οποία θα είναι η βιτρίνα ουσιαστικά των πολιτικών αποφάσεων. Ευχαριστώ κύριε Σικέρσκι. Ευχαριστώ. Πριν από λίγους μήνες είχαμε αποφασίσει να εργαστούμε για τις τροπολογίες για την αγροτική πολιτική χωρίς να τις εξαρτώμε τις αποφάσεις μας από τις αποφάσεις σε θέματα δημοσιονομικών προοπτικών. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τηρήσουμε αυτή την ηλυμένη απόφαση. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε κάποιες πληροφορίες οι οποίες κυκλοφορούν, κάποιες φήμες, ή πληροφορίες σε σχέση με την αλλαγή του δημοσιονομικού πλησίου να μας επηρεάσουν. Για τις τροπολογίες λοιπόν αυτές που έχουμε ενώπιόν μας, να αφήσουμε τελείως στο πλάι όλα αυτά τα θέματα που αφορούν τις πραγματικές ή ενδεχόμενες περικοπές στον προϋπολογισμό. Όταν έχουμε τις τελικές πληροφορίες για τον προϋπολογισμό, τότε μπορούμε να συμπεριλάβουμε αυτά τα σημεία. Επίσης, η έκθεση για τη συνοχή θα αντιμετωπιστεί στην Επιτροπή Περιφερειακών Θεμάτων. Στην Επιτροπή αυτή έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο κλίμα όπου υποστηρίζεται ιδιαίτερα η ενίσχυση της πολιτικής συνοχής. Υπάρχει λοιπόν ένα θετικό ρεύμα υπέρ της συνοχής στην Επιτροπή Περιφερειακών Θεμάτων. Μα <clears throat> η Επιτροπή Περιφερειακών Θεμάτων συγχρόνως βλέπει τη συνοχή ως μια υπόθεση κυρίως των αστικών χώρων. Έχουν ανατραπεί τα πράγματα. Εμείς θέλουμε να υπάρξει μεγαλύτερη αγροτική ανάπτυξη. Το να λάβουμε υπόψη μόνο την ε, διάσταση των, ε, των πόλεων, αυτό σημαίνει ότι μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα οι αγροτικές περιοχές. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να γίνει αυτή η πολιτική συζήτηση από τις πολιτικές μας ομάδες για να έχουμε μια καλύτερη εκτίμηση της πορείας των πραγμάτων και θέλω να σας παροτρύνω προς την κατεύθυνση αυτή. Ουρικ, Ρόδουστ, äh, Παρακολούθησα με μεγάλη προσοχή όλες αυτές τις ε, παρεμβάσεις των συναδέλφων και θέλω να κάνω το εξής σαφές. 2.600 τροπολογίες έχω εγώ στην Επιτροπή Αλίας για τον βασικό κανονισμό και πιστεύω ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια αντίστοιχη κατάσταση στις τροπολογίες για την αγροτική ανάπτυξη και τις άμεσες πληρωμές. Ένα τμήμα των διακοπών μου ήταν να μπορέσω να διαβάσω όλες τις τροπολογίες στον τομέα του βασικού κανονισμού για την αλία. Τώρα, αυτό το οποίο είδα βέβαια είναι ότι πάρα πολλές τροπολογίες είναι ταυτόσιμες, είναι χαλκομανία. Μόνο και μόνο έχουν οι διαφορετικά ονόματα αυτών που τις κατέθεσαν από διαφορετικές ομάδες. Εγώ αντρώ το συμπέρασμα ότι προέρχονται από ομάδες πίεσης, από λόμπι αυτές τις τροπολογίες και απλώς αλλάζουν τα ονόματα αυτών που τις καταθέτουν. Επομένως, τι θέλω να πω. Έχουμε στα χέρια μας την συναπόφαση ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτή τη στιγμή αντί να το χρησιμοποιούμε αυτό βομβαρδίσουμε αυτούς με τροπολογίες οι οποίες εν μέρη επικαλύπτονται και είναι ταυτόσιμες ή αλλάζουν μονάχα σε μία ή δύο λέξεις και τελικά σε επίπεδο ουσίες έχουμε μονάχα καμιά κατοστή τροπολογίες που έχουν πραγματικό ζουμί. Σας παρακαλώ λοιπόν να σκεφτείτε καλύτερα μήπως στο μέλλον θα πρέπει να έχουμε μια καλύτερη αντιμετώπιση ή αν θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή την πορεία η οποία θα μας οδηγήσει σε όλο περισσότερες τροπολογίες, όλο περισσότερες χιλιάδες τροπολογίες. Για τη συζήτηση στις πολιτικές ομάδες μπορώ να πω στη δική μου πολιτική ομάδα ότι τον προηγούμενο μήνα έχουμε συζητήσει, τους προηγούμενους μήνες έχουμε συζητήσει ιδιαίτερα για τα θέματα της αγροτικής μεταρρύθμισης. Θέλουμε μια αγροτική μεταρρύθμιση και ιδίως μια οικολογικού χαρακτήρα μεταρρύθμιση και αυτό είναι ουσιαστικό. Και γι' αυτό δεν νομίζω και σας το λέω αυτό ότι αυτά που λένε οι τροπολογίες είναι κάτι το καινούριο. Οι περισσότερες δεν είναι καινούριες. Το να συζητήσουμε και πάλι όλα αυτά τα πράγματα στις πολιτικές ομάδες, αυτό είναι δύσκολο. Αν δεν το έχουμε κάνει στο παρελθόν, δεν μπορεί κανείς να βγαίνει και να λέει έχω την πρόθεση να προβώ σε μια ουσιαστική μεταρρύθμιση. Είναι πολύ αργά για να περάσουμε σε μια συζήτηση επί της ουσίας πια. Ευχαριστώ, Και εγώ κατάλαβα τα όσα είπε η συνάδελφος Ρόντος. Πιστεύω πως για πρώτη φορά υπήρξε τουλάχιστον είναι προφανής ε, στις ε, τροπολογίες η παρουσία και η συμμετοχή των κυβερνήσεων, πράγμα που Ε, ας πούμε κάποιες τροπολογίες ε, τα, είναι ακριβώς οι ίδιες απο, και υποβλήθηκαν από διάφορες ομάδες. Ε, σίγουρα θα υπάρχουν και λόμπι, αλλά υπάρχουν και ε, κυβερνήσεις που έχουν παρέμβει. Και τώρα θα δώσουμε τώρα το λόγο στον Αντιπρόεδρο Βοσιγόφσκι και μετά θα κλείσει ο Άλμπερτ Ντες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το συγγνώμη που δεν μπορούσα. Ευχαριστώ πολύ. Αφού είναι τόσε πολλές οι τροπολογίε, ας έχουμε το χρόνο να τις επεξεργαστούμε καταλήλω αυτές τι τροπολογίε. να μην ακολουθήσουμε αυτό το μαύρο όραμα, δηλαδή τις περαιτέρω περικοπές ε, των κονδυλίων για τη γεωργική πολιτική. Σαφώς είναι πρόκληση αυτή που πρέπει να αντιμετωπίσει η Γεωργία, η Ευρωπαϊκή Γεωργία και ε, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επιδείξουμε αποφασιστικότητα. Βρισκόμαστε σε πιο δινή θέση σε θέση με τις ε, προοπτικές 2007-2013 και σε ελπίσουμε το τελικό αποτέλεσμα των εργασιών μας για τον προπολογισμό θα είναι τέτοιο ώστε τα κονδύλια της γεωργικής πολιτικής να μην τροποποιηθούν υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, στο οποίο αναφερθήκαμε επανειλημμένως νομίζω, το θέμα της κατανομής των πληρωμών και τις νομικές ε, πτυχές που σχετίζονται με αυτό. Κύριε Πρόεδρε, το έχω ξαναπεί και στο παρελθόν, θα πρέπει να έχουμε τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας για τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται τα κονδύλια. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σέβεται τη συνθήκη. Μπορεί να μην γίνονται σεβαστές οι αρχές της μη διάκρισης μεταξύ των κρατών μελών. Και μπορεί να παραβιάζεται και η αρχή της μη διάκρισης των Ευρωπαίων παραγωγών. Οι πληρωμές θα πρέπει να ε, δίνονται με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν και σαφή κριτήρια που καθαρίζουν τους στόχους με τους οποίους γίνεται κάθε σύγκριση για τις πληρωμές. Για παράδειγμα, ιστορικά κριτήρια δεν αιτιολογούνται. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι ο κάποιος ο οποίος λάμβανε χ ποσοστό χρηματοδότησης πρέπει να λαμβάνει την ίδια χρηματοδότηση. Πρέπει να γίνεται διαφοροποίηση, βεβαίω θα πρέπει να γίνεται διαφοροποίηση, αλλά θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη αιτιολόγηση. Δεν μπορεί να γίνονται αυθαίρετα αυτέ οι διαφοροποίησει. Θα ζητήσω λοιπόν αυτά τα ζητήματα τα νομικής φύσεως ε, να διευκρινιστούν ε, ώστε να έχουμε μια σαφή απάντηση. Και επαναλαμβάνω το αίτημά μου να ληφθεί υπόψη το ζήτημα αυτών και να ζητήσουμε την άποψη των ειδικών. Έχουμε τη δυνατότητα νομικής νομοδότησης. Στο Κοινοβούλιο της Πολωνίας ε, παρουσιάστηκαν ε, σχετικές αναλύσεις που αποδεικνύουν ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν συμμορφούνται προς τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε τον Αντιπρόεδρο, ο Άλμπερτ τώρα. Σας ευχαριστώ. Ζήτησα το λόγο για να πω το εξή ότι έχουμε αυτή τη στιγμή 7.000 και τροπολογίες για τα, τις τέσσερις εκθέσεις. Αυτό δείχνει όμως ότι χρειαζόμαστε και μια μεταρρύθμιση του εσωτερικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ είχα προτείνει στην ομάδα μας ότι η κατάθεση τροπολογιών θα πρέπει να απαιτεί τουλάχιστον 10 υπογραφές συναδέλφων. Αυτό θα μειώσει ριζικά τον αριθμό των τροπολογιών. Πιστεύω ότι πρέπει να συζητήσουμε και για το θέμα αυτό, ώστε τα πράγματα να παραμείνουν στο επίπεδο του λογικού. Αν τώρα η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου δεν είναι διατεθειμένη να ακολουθήσει μια τέτοια κατεύθυνση περιορισμού. μπορεί να φτάσουμε εν καιρό σε 20 με 30 χιλιάδες τροπολογίες, κάτι το οποίο είναι πια αδύνατον να λειτουργήσει. Πρέπει να κάνουμε ότι είναι απαραίτητο να παραμείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα επίπεδα του λογικού, να είναι βιώσιμη και εφικτή η εργασία μας και πρέπει να συζητήσουμε για όλους αυτούς τους λόγους και για την εσωτερική διάταξη των εργασιών μας και τον κανονισμό του Κοινοβουλίου. Ωραία, Albert. Θα συζητήσουμε, Albert. Ίσως στο τέλος αυτής της Επιτροπής να μείνουμε με λίγο με τους συντονιστές και τους εισηγητές, να μιλήσουμε για τη μέθοδο και μετά να ενημερώσουμε και την υπόλοιπη Επιτροπή. Και τώρα θα δίνω το λόγο στην Επιτροπή. Είναι εδώ ο Διευθυντής Πατσέκου και μετά θα δώσω και πάλι το λόγο στον Λουίς. Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω πως αυτό που μπορώ να πω είναι ότι από την πλευρά της Κομισιόν αναμένουμε το Κοινοβούλιο να καταφέρει να λάβει θέση για τις ε, τροπολογίες και είμαστε στη διάθεσή σας, απόλυτη διάθεσή σας, ώστε να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να έχετε βοήθεια βοήθεια και διευκρινήσεις που χρειάζεστε για να φτάσετε, φέρετε σε αίσιο πέρα σε αυτό το τόσο δύσκολο αλλά και σημαντικό έργο. Ευχαριστώ. Ωραία. Ο Λουίς. Κύριε Πρόεδρε, πραγματικότητα είναι αυτή. Δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Άρα πρέπει να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. έχουμε δυνατότητα για μια ευκαιρία για να βρούμε μια καλή λύση για την ε, κοινή γεωρική πολιτική. Όσον αφορά τον καθαρισμό της μεθέδους, φυσικά και είμαστε υπέρ της ε, ε, συνεδρίας των συντονιστών. Το έχω σημειώσει. Όπως είπε η κυρία Μαγκίνες, ίσως καλύτερα είναι να, να ξεκινήσουμε με τα λιγότερο περίπλοκα θέματα. Άλλο συνάδελφος μίλησε για, είπε να ξεκινήσουμε από το greening, το πρασίνισμα. Με πάση περιπτώσει θα πρέπει να καταβάλουμε κάποιες προσπάθειες ώστε να αρχίσουμε να δουλεύουμε γρήγορα. Και φυσικά με μεγάλο ρεαλισμό θα πρέπει να αναλύσουμε όλες τις προτάσεις. Για παράδειγμα, ο συνάδελφος Μαγκίνης μίλησε ε, και, και, και ο συνάδελφος Λάιονς μιλήσαν για το θέμα του μενού ως ένα παράδειγμα ενός θέματος που μπορεί να υπάρξει ε, ε, διαφωνία ανάμεσα στις δικές μου προτάσεις τροπολογίας και τις προτάσεις άλλων ομάδων. Όταν όμως εγώ προτείνω ένα σύστημα οικολογικού, οικολογικής πιστοποίησης το οποίο μπορεί να δίνεται στα κράτη-μελή, δημιουργώ ε, την πιο αποτελεσματικό τρόπο για τη δημιουργία ενός μενού που να μπορεί να το δεχτεί η Κομισιόν. Η Κομισιόν ε, ήταν αδιάλακτη και έχει υποβάλει ένα κατάλογο πολύ εκταμένο για μέτρα greening, πράγμα το οποίο θα αυξήσει το γραφειοκρατικό άχθος θα δυσχεράνει τον, τον έλεγχο και ενώ εγώ πιστεύω πως όταν έχουμε έναν μηχανισμό οικολογικής πιστοποίησης που είναι ένα μέσο το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα κάτι μελη ώστε να γίνουν πιο ευέλικτα τα μέτρα του πρασινίσματος, τότε μπορούμε να βρούμε μια λύση λοιπόν συνενετική και να καλύψουμε τις ανησυχίες όσων δεν θέλουν εξαντλητικό κατάλογο μέτρων, ενώ ταυτόχρονα θα ανταποκριθούμε και στις επιθυμίες εκείνων που επιθυμούν μηχανισμούς ευελιξίας για την εφαρμογή του greening, δηλαδή Δηλαδή θα πρέπει να είμαστε πολύ ευέλικτοι, να, έχουμε πολύ, να επιδείξουμε πνεύμα συμβιβαστικό. Γιατί έτσι αν υπάρχουν δυνατότητες να έχουμε ένα κατάλογο μενού που να μπορούμε εύκολα να τον, ε, τον ελέγξουμε και που θα μπορούν να το εφαρμόσουν οι διάφοροι γεωργοί στα διάφορα κράτη-μέλη, σίγουρα θα βρούμε συμβιβαστική λύση. Στην πράξη βέβαια δεν, δεν είναι και τόσο εύκολο, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει καλή βούληση πιστεύω ότι δεν υπάρχουν ε, ανεπίλητα προβλήματα. Θα πρέπει λοιπόν να επιδείξουμε ρεαλισμό και βούληση και παρά τη δυσκολία είμαι αισιόδοξο όσον αφορά την έκβαση των εργασιών μας. Σα ευχαριστώ συνάδελφοι, ευχαριστώ, ευχαριστώ για τη συζήτηση και τώρα λοιπόν θα οργανωθούμε. Σίγουρα η γραμματεία θα μας βοηθήσει στο να συστηματικοποιήσουμε αυτή την μάζα τροπολογιών όπως φαντάζομαι εξάλλου και σε αυτή την πρώτη συνεδρίαση των συντονιστών που θα κάνουμε και των εισηγητών θα θέσουμε κάποια κριτήρια. Η ευθύνη είναι μεγάλη, πραγματικά πολύ μεγάλη. Καλούμαστε, ως κοινοβούλιο να ε, συμβάλλουμε ε, ώστε να γίνει μια καλή μεταρρύθμιση σύμφωνα με την συνθήκη της Λισαβόνας και τη συναπόφαση και όχι μια μεταρρύθμιση πάση θυσία, αλλά μια μεταρρύθμιση που θα δώσει απαντήσεις στα προβλήματα. Να σας θυμίσω λοιπόν, οι επόμενες συνεδριάσεις έχουν οριστεί για τις 17 ε, Σεπτεμβρίου στις 3 ε, και στις 7 Σεπτεμβρίου κλείνει τώρα τέλος της συνεδρίας αυτής. Θα μείνουμε 5-10 λεπτά και ζητώ από τους συντονιστές και τους συζητητές να μείνουν στην αίθουσα. Ευχαριστώ.